τον κύριο Γύρι Μαστάλκα και τον κύριο Ρίκο Περόνι τους όρισα ως ε, αναπληρωτές ε, από τους ομάδες του ΕΛΚ, του ΑΛΔΕ, των Πρασίνων και της ΓΚΟΥΝΕ και των μη Έλαβα ε, υποψηφίους και ο κατάλογος θα δημοσιευτεί στα πρακτικά. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι γίνονται αυτές, αυτοί οι διορισμοί να σας ανακοινήσω ένα